cominciamo. Buonasera a tutti. Allora, chiesto velocemente la parola l'onorevole Audi. Prego. Ο κύριο Οντί έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη να επανέλθω σε ένα απονεμένο σχέδιο για το 108 του κανονισμού για το διορισμό του κυρίου Φαζάκα. Θα ήθελα να ξέρω με ποιο καθεστώς θα πάει αυτό το έγγραφο στην Ολομέλεια. Φαίνεται να είναι έκθεση του ελέγχου του προπολογισμού. Η συνάδελφος Αγιάλα Σέντερ έκανε εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν ψηφίσαμε όμως εμείς για αυτή την έκθεση. Για, τα, για το όνομα ψηφίσαμε, για την έκθεση δεν ψηφίσαμε. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο αυτό το έγγραφο έχει κάποιο συγκεκριμένο καθεστώς. Τι είναι. Αν περάσει ως έκθεση δηλαδή το ελέγχο του προϋπολογισμού, εμείς δεν το ψηφίσαμε. Και από τώρα και μέχρι την ε, Ολομέλεια θα πρέπει, ε, ε, θα μπορέσουν βάσει του άρθρου 108 να ζητήσουν και αναβολή. Εμείς είχαμε απάντηση της Ουγγαρέζικης κυβέρνησης, αλλά δεν απαντάει στο ζήτημα. Αυτό το οποίο μας απασχολεί εμάς ως βουλευτές είναι ότι ο κύριος Φαζάκα είπε ψέματα. Λοιπόν, ε, εμείς δεν μπορούμε να διορίσουμε στο ελεγκτικό συνέδριο κάποιον που λέει ψέματα. Είτε ο κύριος Ντόιτς λέει ψέματα, είτε ο κύριος Φαζάκα. Και τελικά η Ουγγρική κυβέρνηση δεν μας το είπε. Μας λέει ότι ο κύριος Φαζάκα έχει ένα δεύτερο όνομα. Λοιπόν, δεύτερο όνομα τι όνομα, όπως ισχύει σε ορισμένες χώρες που έχει κάποιος δύο ονόματα ή στην περίπτωση του κυρίου Φαζάκα είναι ένα όνομα δίπλα το οποίο είναι κωδικό. Λοιπόν, μπορούμε εμείς να ενημερώσουμε την Ολομέλεια για όλες τις απορίες που έχουμε και να διαφωτίσουμε και τους συναδέλφους μας όταν έρθει η ώρα στην Ολομέλεια. Κύριος Μπρέγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι κρίμα να ασχολούμαστε τώρα με αυτό, γιατί εγώ θεωρούσα ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία που ανέφερα και στους συντονιστές. Το λέω και για την ομάδα και για την Επιτροπή. Όσοι είναι πιο πολύ καιρό εδώ στην Επιτροπή να πω καταρχάς ότι δεν είναι η πρώτη περίπτωση όπου διάφοροι αμφισβητούνται διάφοροι αξιωματούχοι κυβερνήσεων ανατολικών χωρών. Κατά δεύτερον, στην προηγούμενη οφαντική περίοδο η Επιτροπή δικαίως περιορίστηκε στα καθήκοντά της. Δεν ε, έλεγξε ως δικαστήριο τη λειτουργία των ε, αξιωματούχων αυτών, απλά κοίταξε όσα εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της. Εγώ πολύ απλά, κυρία Όντι, θα ήθελα να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, επειδή υπάρχει και, υπάρχει και απόφαση της Επιτροπής και της Ολομέλειας εμείς λοιπόν έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας και η επιστολή αυτή δεν ε, έχει καμία τέτοια σάφια. Ε, Εγώ θέλω να προσθέσω το εξή. Εχθές στους συντονιστές αποφασίσαμε να συζητήσουμε στην ημερήσια διάταξη το πώς θα συμπεριφέρεται κανονικά, δηλαδή ένας κώδικα συμπεριφοράς της Επιτροπής μας, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή αυτό το οποίο συνέβη τις προάλλες για το διορισμό του Φαζάκας, ε, αν μας συμβεί μια άλλη φορά πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε. Τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς είχαμε μια ψηφοφορία η οποία έδωσε μία ένδειξη σαφή προς την Ολομέλεια σχετικά με τον Φαζάκας. Ότι θα έπρεπε δηλαδή να σταλούνε από την Ουγγρική κυβέρνηση για να ξέρουμε να μας πει τι ακριβώς έγινε, ποια ήταν η ψηφοφορία, πώς ψηφίσαμε την επιστολή του Υπουργού από την Ουγγαρία και μετά οι διάφορες πολιτικές ομάδες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον διορισμό του Φαζάκας. Εγώ δίνω το λόγο στον Ντόιτς, παρακαλώ όμως να είμαστε σύντομοι γιατί αυτό το θέμα δεν είναι στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να ψηφίσουμε. Ο κύριος Ντόιτς, σύντομα. Αμάν. Σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση αυτή. Και θεωρώ ότι το θέμα αυτό το οποίο έφυξε ο κύριος Οντή, ο Αντιπρόεδρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και θεωρώ ότι δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Όντι από τον Πρόεδρο. Να προσθέσω το εξή κύριε Πρόεδρε. πάντα έχετε θίξει θέματα της Ουγγρικής ε, κυβέρνησης και σας έδωσε ε, απάντηση η Ουγγρική κυβέρνηση. Έχετε λοιπόν την ε, σαφή απάντηση της Ουγγρικής κυβέρνησης η οποία περιέχει ένα σαφές ψέμα. Αυτό το ψέμα κορεδεύει όχι μόνο όλη την Επιτροπή αλλά και όλο το Κοινοβούλιο. Στην απάντηση που έδωσε η Ουγγρική κυβέρνηση αναφέρεται ότι ο κύριος Φόσακος ότι υπάρχει έγγραφο από το Υπουργείο Ιστορικών. Το έγγραφο όμως που σας δείχνω αυτή τη στιγμή είναι η χάρτα υπαρθμών έξι του κυρίου Κόσακος όπως αποκαλείται. Αυτό αποτελεί ένα ένα ψευδόνυμο το οποίο χρησιμοποιούσε παλαιότερα. Όχι Στέφαν. Μιλάμε για σαφές ψέμα της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης και κάπως θα πρέπει να αντιδράσει η Επιτροπή μας. Ναι, συμφωνώ ότι δεν, θα, δεν είμαστε δικαστήριο, αλλά και ένα δεκάχρονο παιδί μπορεί να ξεχωρίσει το ψέμα αυτό το πασιφανές. Όποιος έχει μάτια και διαβάζει, βλέπει αυτό το ψευδόνυμο, το Στέφαν, αλλά η Ουγγρική κυβέρνηση τώρα βγαίνει και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για το δεύτερο όνομά του. Δεν ισχύει αυτό. Ως Στέφαν αναφέρεται στα αρχεία της ε, των μυστικών υπηρεσιών της Ουγγαρίας. Καταλαβαίνουμε την πρόταση φυσικά που έγινε και καταλαβαίνω ότι κάθε ομάδα θα διαμορφώσει τη δική της τοποθέτηση, αλλά παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα στοιχεία αυτά, να ενημερωθούμε γραπτά προκειμένου και οι ομάδες και οι βουλευτές να μπορέσουν να αποφανθούν. Ε, ναι. Η κυρία Γκρέσλε, πολύ φοβάμαι ότι με, μετά από αυτή την συζήτηση θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν. Δεν μπορούμε ούτε πρέπει να αποφασίσουμε, ούτε μπορώ να κρίνω και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περάσουμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Ε, Ωραία, συνεχίζουμε. Γιατί αν, ε, αντίθετα από αυτό που είπε ο κύριος Δόιτς εγώ ανταποκρίθηκα ε, προηγουμένως απαντώντας σας δηλαδή για τα ζητήματα ελέγχου. Λοιπόν, ας ε, προχωρήσουμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε. Μπορούμε αν θέλετε να το συζητήσουμε στο τέλος της συνεδρίασης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, μίλησα για αυτό το θέμα στη συνεδρίαση των συντονιστών και θα, ήθελα να ρωτήσω ποιος εκπροσωπεί το ΕΛΚ, η κυρία Γκρέσλε ή ο κύριος Ντόιτς. Έχω την εντύπωση ότι όλοι ανήκουν και οι δύο ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα. Ε, μήπως έχουν αλλάξει κανόνες και δεν το ξέρω. Το... Ναι, Συγγνώμη, στην Επιτροπή του Ελέγχου του Προπολογισμού ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του και έχει δικαίωμα να μιλάει. Λοιπόν, η κυρία Γκρέσλερ είναι συντονίστρια του ΕΛΚΑ. Λοιπόν, η κατάσταση είναι σαφής, εγώ λέω να προχωρήσουμε και μετά άμα έχουμε χρόνο μπορούμε να ξανασυζητήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Απαλλαγή 2008, Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα 3, Επιτροπή. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Λιμπεράτσκι, θέλω να χαιρετήσω τον Ατζίλντα Σεμέτα, τον Επίτροπο που είναι παρόν και θέλει να κάνει μία δήλωση. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Η, απαλλαγή, διαδικασία απαλλαγή του 2008 είναι σε προκεχωρημένο στάδιο. Ε, ήταν εντατική η ρυθμή και κυρίως ξεκίνησε ένας νέος διάλογος. Ε, Είχα έρθει με τους συναδέλφους μου για να σας περιγράψω την κατάσταση και να σας μιλήσω για τις μελλοντικέ προοπτικές ε, στον πλέον κρίσιμο τομέα των διαρθρωτικών ε, ταμείων. Έχετε λάβει μία ε, επιστολή του κυρίου Λεβαντόφσκη και μου του ίδιου σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό. Με τον κύριο Σεύκοβιτς σας έστειλα ένα κατάλογο των μη μικρών που λαμβάνουν νοσιακή χρηματοδότηση. Φυσικά θα εξετάσω ε, με προσοχή τις συστάσεις του Κοινοβουλίου τον Απρίλιο και θα ε, εξασφαλίσω θα υπάρξει σωστή συνέχεια. Αυτά είναι τα πρώτα βήματα που καταδεικνύουν την ισχυρή δέσμευση και αφοσίωσή μου για συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ενώ ταυτόχρονα οι συνάδελφοι επίτροποι θα εμπλακούν εξίσου ενεργά στη διαδικασία. Θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν ε, να αναβαθμίσουμε τις δαπάνες ε, ως προς την ποιότητα τους δηλαδή και θα συνεχιστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη. Φυσικά επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση η κατάσταση. Η απλουστευμένη νομοθεσία και τα διάφορα σχέδια δράσης κοινή διαχείριση δείχνουν ότι υπάρχει ένα ασθετικός αντίκτυπος ως προς τα ποσοστά λάθους. Ε, και αναμένουμε ότι τα πρώτα αυτά αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται από το φετινό δημοσιονομικό έτος. 2010 και εξής δηλαδή. Ταχεία προόδο όμω είναι αδύνατη αν δεν συμμετέχουν ενεργά και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορεί και τα κρατημέλη και φυσικά το ελεγκτικό συνέδριο. Χρειαζόμαστε ενεργό εμπλοκή των κρατών μελών για να επιτύχουμε τους στόχους μας ταχύτατα. Με του συναδέλφου επιτρόπου, δεν θα περιμένουμε την τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, δεν περιμένουν να αρχίσουν να ισχύουν. Καλούμε ήδη τι εθνικέ αρχέ να υπομιστούν τι ευθύνε του σε βάση τη τη Λισαβόνα και περιμένουμε να υλοποιηθούν τα μέτρα που θα αναβαθμίσουν τη δημοσιονομική διαχείριση. Θεωρώ επίσης ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο ούτως ώστε ε, να ε, εξασφαλιστεί χρηστή οικονομική διαχείριση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, οι προϊούσε συζητήσει του ελεγκτικού συνεδρίου και οποιασδήποτε αλλαγές θα γίνουν ε, φυσικά θα συνεπάγονται, θα επισύρουν και άλλες αλλαγές ως προς τα ποσοστά ε, λαθών. Ε, ως προς τους τομείς τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Παραδείγματος χάρη ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα προγραμματική περίοδο όταν ε, ο συνομοθέτης ε, θα συμφωνήσει σχετικά με το ανεκτό ποσοστό λάθος, ελπίζω, λάθος, ελπίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο τελικά θα εγκρίνει αυτά τα πορίσματα. Όπως ζήτησε η Επιτροπή, θα σας παρουσιάσω το Μάιο χρονοδιάγραμμα απαλλαγής ε, ελέγχου και μέτρων καταπολέμησης απάτης για τα επόμενα έτη. Η εμπλοκή όλων των εταίρων με κοινό στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων τη Ευρωπαϊκής Ένωση, θα είναι στον πυρήνα αυτού του προγράμματο που θα σας παρουσιάσω το Μάιο. Συνοψίζοντας, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λιμπεράτσχη, τον εισηγητή σας. Εργάστηκε σκληρά για την απαλλαγή του 2008 ε, και με μέλη, να ευχαριστήσω και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ε, για τη συνεργασία τους, την υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσουμε την οικονομική διαχείριση και την εκτέλεση του νοσιακού προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο Σεμέτα. Τώρα ο κύριος ε, και ο εισηγητής μας. <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να μιλήσω για την έκθεση αυτή. Η διαδικασία χορήγηση απαλλαγή είναι πάντα ένα περίεργο μείγμα. κοιτάμε προ τα πίσω και κοιτάμε και προ τα μπροστά. Και αυτή η φορά δεν ε, αποτελεί εξαίρεση. Βρισκόμαστε στην φάση εκκίνηση μια νέα επιτροπή και θα πρέπει να υπερβούμε τα προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε από προηγούμενα προγράμματα. Είμαστε Είμαι ευγνώμων για την ε, συμβολή πολλών συναδέλφων της Επιτροπής μας ε, από τους Επιτρόπους και το προσωπικό της Επιτροπής και τη συμβολή όλων ε, των μελών της Γραμματείας της Επιτροπής που εργάστηκε πολύ σκληρά. Προσπάθησα να ισορροπήσω, να εξορροπήσω την κριτική για αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν με κάποια στοιχεία και προτάσεις για το μέλλον, γιατί η νέα συνθήκη δίνει έμφαση στην κοινή ευθύνη των κρατών μελών με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σε ό,τι αφορά την διαχείριση των προπολογισμών. Επίσης αναφέρονται σημαντικά βήματα τα οποία θα πρέπει να αναλευθούν σε διάφορα επίπεδα. Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική. Το τονίζω αυτό, δεν είναι ικανοποιητική. Και γι' αυτό το λόγο συμπεριέλαβα την έκκληση να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να γίνει προσπάθεια να προσεγγίσει το χρονοδιάγραμμα αυτό την περίοδο που αναφέρεται, στην οποία αναφέρεται ε, η απαλλαγή. Καταλαβαίνω ότι πρακτικά προβλήματα μπορούν να ε, προκληθούν και έχω θέσει και στόχους για τις ε, βελτιώσεις οι οποίες θα πρέπει να συμβούν και Αυτά λαμβάνονται σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θεωρώ ότι οι στόχοι αυτοί έχουν ήδη ε, ληφθεί σοβαρά υπόψη από την τρέχουσα Επιτροπή. Επίσης, ε, στην έκθεση ζητώ από το δικαστήριο να μας δώσει τη δυνατότητα για πιο λεπτομερή ανάλυση της απόδυσης εντός της πολιτικής συνοχής ακόμα και με ξεχωριστή ανάλυση των διαφόρων τομέων προγραμμάτων ή με διαφορετικές διαδικασίες για άσκηση ελέγχου για την παλιά και την καινούργια νομοθετική περίοδο. Ανυπομονώ και ελπίζω στη συνεργασία σας και την υποστήριξή σας και εδώ και στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια όλου του follow-up. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Λιμπεράσκη, για τη δουλειά του. Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Απαλλαγή λοιπόν στον προπολογισμό για την Κομισιόν το 2008. Ψηφίζουμε την πρόταση για την απαλλαγή στο σύνολό της, η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τα σημεία 1 ως 4, αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνονται 24-4 Η πρόταση στο σύνολό της αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε για τα όπτικα οπτικακουστικά, για την απαλλαγή αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25-4. για τον ανταγωνισμό και την καινοτομία. Α, ένα λεπτό. Πάμε πίσω. Λοιπόν, για το οπτικά ακουστικά και τον πολιτισμό. Λοιπόν, ψηφίζουμε την πρόταση στο σύνολό της. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην απαλλαγή ε, στον εκτελεστικό οργανισμό για τον ανταγωνισμό. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Πρόταση στο σύνολό της. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες. Ε, οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές. Ε, ψηφίζουμε. πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 25-4. Πρόταση ούτως τροποποιημένη. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίες, Εγκρίνεται. Λοιπόν, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. 23-4. Πρόταση στο σύνολό τη. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών με αναφορές στα σημεία 14, 15, 16, 17. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 24-4 λοιπόν. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 19. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τελική πρόταση, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24-4 πρόταση ψηφίσματος. Προφορική τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 20. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 22. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 23. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αποσύρθηκε 24-25. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 27. 28. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Το 30, το 30 πρέπει να ψηφίσουμε. Ωραία, λοιπόν, 30. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 32. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 33 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Προφορική τροπολογία 3 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 35 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες Εγκρίνεται. 36. Αρχής ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίας. 37. αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 39. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 40. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σαρανταένα, Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 42. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Unblock. Τροπολογία 43 ως 45. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 48. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 49. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 50. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. εγκρίνεται. 52. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 53. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 58. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 60. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 61. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 62. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέρες ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5 αρχίζει ψηφοφορία. Τέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 64. Αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 65. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 66. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 68. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 69. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 70 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. δύο αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. τέσσερα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 73 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες εγκρίνεται. Η προφορική τροπολογία 6 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρες ψηφοφορίες εγκρίνεται. 76. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 77. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 78. Απορρίφθηκε. 80. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 81. Πέρας ψηφοφορίας. 83. Πέρασε εγκρίνεται. 84 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. 85 αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 86 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε Εγκρίνεται. 87. Απορρίφθηκε. 88 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 89. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 90. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 91. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε. 92 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. ψηφίζουμε 94-95-96 Πέρασε. Απορρίπτεται. «97 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία». Τέλος. Απορρίπτεται. Το δεύτερο τμήμα της 97. Αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 98 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 99. Α, όχι, έχει καταπέσει. 100. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 102 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 103 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 104 Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 105. Αρχή ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 107. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 108 αρχίζει ψηφοφορία πέρας της. Ψηφοφορίες εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7. Εγκρίνεται. 110. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Προφορική τροπολογία 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 113. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 114. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 115 σε τρία χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 116. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 118. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 9. Κύριε κύριος Γκρέι. Συνάδελφοι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να κάνω μια προφορική τροπολογία. Θα ήθελα εκεί που λέει στο staff regulation να αναφέρω τη λέξη στα αγγλικά. Αμφισβητεί την ε, εφαρμογή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφέρεται contest στα αγγλικά. Θα ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο έντονο, να πούμε deplores. Ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία ούτως τροποποιημένη από τον κύριο Γκρέιερ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 120 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 121 αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 122 χωριστό, χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. 123 Πέρας. ψηφοφορία εγκρίνεται. 124. Εγκρίνεται. 125. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 126. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 10. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 128. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 11. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν τριάντα και εκατόν τριάντα ένα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η πρώτη της περιφερειακής αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 133 αρχίζει η ψηφοφορία. 132, συγγνώμη, μπερδεύτηκε. λοιπόν. 132. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 134 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 135 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 137. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 138. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 9 της Περιφερειακής. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 139. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 12. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δέκα της Ρέτζη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρία της Ρέτζη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας Φώτιας. Προφορική τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 140. Ε, Πέρασε. Εγκρίνεται. 141 αρχίζει ψηφοφορία. Εκατό σαράντα δύο. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Οχτώ της Ρέτζη. Αρχίζει ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται. 5 της Ρέτζη αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6 της Ρέτζη. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 143. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. εφτά της Ρέτζη. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 144. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 145 πρώτο τμήμα Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 της Ρέτζη. Εγκρίνεται. 12. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13 της Ρέτζη αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γνωμοδότηση 1. Ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 3. Πέρασε. Απορρίπτεται. από τη γνωμοδότηση απασχόληση από το 4 μέχρι το 10 μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ. Αρχίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 146 ψηφίζουμε. Πέρας τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 147 ψηφίζουμε. Πέρας τις ψηφοφορίες φορές. Απορρίπτεται. 148. Εγκρίνεται. 149. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 150. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας Δεν Εγκρίνεται. Από το 1 ως 8 ψηφίζουμε έναν μπλοκ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εννέα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ένα ΙΜΚΟ. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 2. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 3 ως 5. Ψηφίζουμε, unblock. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ίμκο 6, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Από το 1 μέχρι το 11 μπορούμε να ψηφίσουμε unblock. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το 12 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Λοιπόν, Επιτροπή Πολιτισμού, ένα. Πέρας ψηφοφορία. Δύο. Ψηφίζουμε. Πέρας πληροφορίες. Εγκρίνεται. Τρία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Τέσσερα αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, εγκρίνεται. Πέντε αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, Εγκρίνεται. Έξι αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, Εγκρίνεται. Εφτά. Αρχίζει η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Οχτώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εννιά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δέκα. Απορρίπτεται. Λίμπε 1 με 3 αμπλοκ. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αμπλοκ 151-157. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Γυναίκες 1 μέχρι ανάπτυξη 10 αμπλοκ. Πέρα ψηφοφορίες εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία αριθμό 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 15. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 160 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 16 προφορική τροπολογία αρχίζει ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 162 ψηφίζουμε απορρίπτεται. Η 162. Προφορική τροπολογία 17. Πέρας της, τροπο... της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. 165. 166 ψηφίσμα. Πέρας Δεν Εγκρίνεται. 167. Απορρίπτεται. 168.

Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα δύο. Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα τρία. Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα τέσσερα. εγκρίνεται. 170, συγγνώμη, προφορική τροπολογία 18. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 176 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 177 το πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 178. Εγκρίνεται. 179 εγκρίνεται 180 αρχίζει η ψηφοφορία εγκρίνεται 181 αρχίζει η ψηφοφορία πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται

189-190 μαζί ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αρχίζει 191. Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Εκατόν τέσσερα. Εκατόν ενενήντα πέντε. Εγκρίνεται. Εκατόν ενενήντα έξι. 196 Πέρσι, εγκρίνεται. 197 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρσι ψηφοφορία, εγκρίνεται. 198 αρχίζει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Άφετ 5. Όχι, όχι, έχει καταπέσει. 199. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 200. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 201. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 202. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 203. Πέρας απορρίπτεται. 204. Απορρίπτεται. 205. Πέρας Εγκρίνεται. 206. εγκρίνεται. 207. Εγκρίνεται. 208. Αυτό έχει καταπέσει λοιπόν. Τώρα. Τελική ψηφοφορία στο σύνολό της, στη σωστό σύνολο του ψηφίσματος, πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ και 4 κατά και μία από εκεί. Ευχαριστούμε κύριε Λιμπεράσκη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, Έχουμε την απαλλαγή 2008 των άλλων θεσμικών οργάνων. Ο κύριος Τσαρνέκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έβγαλα το σακάκι μου γιατί κάθε φορά με πιάνουν κάποιες κάψες, λέει ο μιλητής, όταν μιλώ για τον προϋπολογισμό. Ε, πριν από λίγες εβδομάδες ε, κάναμε τελική συζήτηση για αυτό το θέμα και έχουν ε, υποβληθεί εκ τότε πολύ σημαντικές τροπολογίες. για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Συμβούλιο και για άλλα θεσμικά όργανα και για να μην πολυλογώ, θα συνοψίσω λέγοντας ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το Συμβούλιο, δεν είναι καινοφανές, το είχαμε και πέρσι. Και τελικά τον Νοέμβριο εγκρίναμε την απαλλαγή για το Συμβούλιο. Αυτή τη φορά, Πρόεδρε, συναντηθήκαμε με ειδικού εκπροσώπους του Συμβουλίου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση, αλλά δεν επαρκεί όμως. Μας διαβίβασε έγγραφα το Συμβούλιο, τα οποία παρουσιάζουν επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. αλλά δεν καλύπτουν όλη την περίοδο, το 2008 δηλαδή, αναφέρονται στο 2007. Εγώ έχω σπουδάσει ιστορία και από ιστορικής πλευράς με ενδιαφέρουν τα έγγραφα που μας έδωσε το Σύμβουλο, αλλά ουδέμια σχέση έχουν με το οικονομικό έτος που εξετάζουμε και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να χορηγήσουμε απαλλαγή για το 2008 ως εκ τούτου. Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να ε, θεωρούμε θα εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ισότιμη εταίροι του Συμβουλίου. Αποταδίκαμε λοιπόν στο Συμβούλιο για να μας διαβάσει και άλλα έγγραφα, αλλά δεν τα λάβαμε. Κρίνω λοιπόν πως σήμερα δεν πρέπει να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Το θέμα θα παραμένει ανοιχτό αν συμφωνήσετε μαζί μου. Περιμένουμε νέες προτάσεις από πλευρά Συμβουλίου, αλλά είναι πρόωρο να χορηγήσουμε σήμερα απαλλαγή. Αυτό προτείνω στα μέλη της Επιτροπής μας. Για τα λοιπά όργανα, έχω δεχθεί ουσιαστικά όλες τις τροπολογίες. Εάν διαπιστώσετε δεν συμπεριέλαβα κάποιες από αυτές τις τροπολογίες, αυτό σημαίνει ότι τις ενσωμάτωσα σε άλλες τροπολογίες που γενικά έγιναν δεκτές. Και θεωρώ ότι έχει βελτιωθεί η Λίανη έκθεση σε σχέση με την αρχική πρόταση που υπέβαλα στην Επιτροπή. Ε, ευχαριστώ τους συντονιστές και ευχαριστώ όλους τους συντάκτες τροπολογιών. Όλοι εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Πρόεδρος, περνούμε τότε στην ψηφοφόρια. Α, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ε, ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς τα σχόλια του Συμβουλίου. Θα ήθελα πριν από την ψηφοφορία να ακούσουμε και κάποια σχόλια από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου ή δυνατόν. Μα ε. Είναι εδώ κανείς από το Συμβούλιο που θέλει το λόγο που μπορεί να μιλήσει δηλαδή μετά από το αίτημα του κυρίου Σόντερ. Ουδής. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1 για την γενική απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 26 κατά μία ψήφος υπέρ. Proponiamo adesso, eh, votiamo il rinvio del discarico dai punti 2 al punto 5. la Ψηφίζουμε τώρα τα σημεία 2 έως και 5. Αρχίζει η ψηφοφορία για την αναβολή της απαλλαγής. Πέρας. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Τώρα, ε, τελική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Πάμε στο σχέδιο ψηφίσματος, τροπολογία υπαριθμών 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία σε. Σι, στα αγγλικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Θα μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε με την τροπολογία που φέρει το, το γράμμα ε, λατινικού αλφαβήτου D. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11 τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία, το γράμμα ε. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 16. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία φέρει το γράμμα 7. F, συγγνώμη. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Να τα ψηφίσουμε ομαδών. Ομαδών λοιπόν τα γράμματα α, β και g. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 21. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 22. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 23 και 24. Αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Άρχεται η τελική ψηφοφορία για το σχέδιο. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή μας. Απαλλαγή για το δικαστήριο τώρα. Ε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το σχέδιο στο σύνολό του. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ε, ψήφους υπέρ και μία κατά. Τροπολογία 1 υπέρ. Ε, συγγνώμη, ε, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο στο σύνολό του. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ. Τώρα, περνάμε στην απαλλαγή του ελεγκτικού συνεδρίου. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, μία κατά. Τώρα για την πρόταση στο σύνολό της αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο στο σύνολό του τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 27 ψήφους υπέρ και μία κατά. Τώρα, περνούμε στην ψηφοφορία για την απαλλαγή για την ΕΟ και Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Τώρα το, την πρόταση στο σύνολό της αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο στο σύνολό του. Αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους ε, υπέρ και 2 κατά. Τώρα περνάμε στην απολογή, απαλλαγή για την Επιτροπή των Περιφερειών. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε με 25 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο στο σύνολό του, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία με το γράμμα Α. Προφορική τροπολογία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Αρχίζει ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Αρχίζει ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Το ψήφισμα στο σύνολό του τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Θα περάσουμε τώρα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρώτα απ' όλα την απαλλαγή. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ. Θα ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο στο σύνολό του. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε με 29 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια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 Ζητώ συγγνώμη γιατί μου ξέφυγε ένα. Έχουμε να ψηφίσουμε και για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Παρακαλώ για την απαλλαγή. Ψηφίστε. Πέρας. 28 ψήφοι υπέρ. Εγκρίθηκε. Τώρα το σχέδιο στο σύνολό του. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 28 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή, εγκρίθηκε. Ψηφίστε το σχέδιο στο σύνολό του. Παρακαλώ, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Perfetto. Complimenti. Τελεία συγχαρητήρια. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων κατά πολέμηση της απάτης ετήσια έκθεση 2008. Δίνω το λόγο στον κύριο Κοτσολίνο. Allora, ε, Συντομότατος θα είμαι. Στην έκθεσή μου τονίζονται τα καυτά σημεία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης. Λαμβάνω υπόψη τις συνεισφορές όλων των συναδέλφων, γι' αυτό η τελική μου έκθεση είναι πολύ πιο πλούσια από αυτή που είχαμε παρουσιάσει στην αρχή. 36 τροπολογίες είχαμε, και είχαμε υποδείξεις και από την Περιφερειακή Επιτροπή. Αποτέλεσμα. Δέκα συμβιβαστικές τροπολογίες, μία προφορική του εισηγητή και μία voting list όπου οι περισσότερες ε, τροπολογίες έχουν ενσωματωθεί. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες επικεντρώθηκαν κυρίως γύρω από τέσσερα σημεία. Αποτελεσματικότητα των ελέγχων, δηλαδή τη δαπάνη των κρατών μελών γι' αυτό, μείωση των παρατυπιών βελτιώνοντας τους κανονισμούς που θα έχουν διαφανείς εφαρμοστικές λεπτομέρειες, κατά πολέμηση της, ε, των καταχρήσεων, διαφάνεια και υγιείς δημοπρασίες, Όλαφ, λειτουργική ανεξαρτησία της Όλαφ, τα κενά στη συνεργασία με, τα κράτη-μέλη και τα προβλήματα που έχει η Όλαφ στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Είχαμε μία διαφορά δε ανατολισμού με έναν συνάδελφο σχετικά με την προσαρμογή του ανθρωπίνου δυναμικού της Όλαφ αν το απαιτήσει νέα στρατηγική. Επίσης, αποφασίσαμε να έχουμε σαφή αναφορά στις χώρες εκείνες όπου γίνονται αυτές οι παρατυπίες. Αυτό είναι μια παλιά παράδοση εξάλλου του Κοινοβουλίου, να λέει τα σίκα σίκα. Εγώ λοιπόν είμαι ικανοποιημένος από τη δουλειά που κάναμε για τη συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και πιστεύω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε θετικά τις εργασίες μας σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε. Τροπολογία 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 2. Ε, μάλλον, συγγνώμη, εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε, με την Περιφερειακή Επιτροπή. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 9 της Ρέτζη. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 7 αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Απόφαση συμβιβασμού 8. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Αποσύρθηκε η 8. Πάμε στον συμβιβασμό 9. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 10. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Συμβιβασμός 10. αρχή φορή. Πέρας ψηφοφορίας. Συμβιβασμός 2. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 το δεύτερο τμήμα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22. Εγκρίνεται. 23. Πρώτο τμήμα. Αρχής ψηφοφορία. Δεφ, ε, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Εγκρίνεται. 24. Εγκρίνεται. 26. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Αρχή ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Ψηφίζουμε. εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 πέρες ψηφοφορίες εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 27 ψηφίζουμε πέρες ψηφοφορίες εγκρίνεται. 28 Έγκρινεται. 29 αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31 αρχή ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 32 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβασμός 6 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβασμός 7 εγκρίνεται 35 Αρχής ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε στο σύνολό της την έκθεση. Ψηφίζουμε. Πέρας τις ψηφοφορίες εγκρίνεται 25 υπέρ, 2 αποχές, συγχαρητήρια κύριε Κοτσολίνε. Τελειώσαμε. Στις 25 Μαρτίου δεν έχει συνεδρίαση. 26 Απριλίου θα συνεδριάσουμε. Στις 3. Καλό απόγευμα. Αμήν.